Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? First of all, can I ask you to... Λοιπόν, συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε και να εγκρίνουμε αμέσως την ημερήσια διάταξη. Αν συμφωνείτε. Καθώς και τα πρακτικά τα πρακτικά της ε, συνεδρίας της 6 Σεπτεμβρίου και το συνεδρίασης της 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Συμφωνείτε? Ωραία, ευχαριστώ. Επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη είναι η απλοποίηση της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων. Είναι ένα σχέδιο γνωμοδότησης από τον κύριο Πέρκερ. Πίρκερ. Έχετε το λόγο. Danke, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Προσπαθήσω να λύσω κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα και δεν σας άκουσα και παρακαλώ να με συμπαθάτε. Είναι σημαντική τούτη εδώ η πρόταση, πιστεύω, προ όφελο των ενδιαφερομένων και των ενεχομένων είναι απλούστευση της Ε, μεταφορά στο εσωτερικό της ενιαία αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτο μέλο. Επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή εσωτερική αγορά Δεν γνωρίζουμε ακόμα το δικό του χρονοδιάγραμμα για την ψηφοφορία. Εμεί όμω αξιοποιήσαμε την ευκαιρία εγκαίρω να κάνουμε γνωμοδότηση από πλευρά τη επιτροπή Μεταφορών. Τονίζω μερικά σημεία, τα έχω σημειώσει για να επανέλθω. Και να πω ότι έχουμε και χρόνο για τροπολογίες μέχρι 16 Νοεμβρίου. Οπότε μπορούμε να κάνουμε την ισχύα μας στις συζητήσεις. Καταρχάς θα ήθελα σύντομα να εξηγήσω τα βασικά σημεία και τους στόχους του κανονισμού αυτού. Και μετά πάλι σύντομα να έρθω στα σημαντικότερα σημεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πω ότι ε, πρέπει εμείς να αντιπροτείνουμε στη γνωμοδότησή μας, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, ε, ως άποψη της Επιτροπής Μεταφόρων. Πρώτον, να κοιτάξουμε τους στόχους. Ποιοι είναι αυτοί. Η ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση οχήματα που έχουν ήδη ταξινομηθεί σε ένα κράτος μέλος. Να υπάρχει τέτοια δυνατότητα και να είναι και πραγματικότητα. Αυτό είναι σημαντικό, ας πούμε, για κάποια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που αγοράζει κάποιος σε μια χώρα και μετακομίζει ή όταν αλλάζει τόπο κατοικίας ή αν μένει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διαμένει σε κάποια άλλη χώρα. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα κάποιοι εργαζόμενοι που για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα πηγαίνουν να εργαστούν σε άλλη χώρα και θα πάρουν μαζί του το αυτοκίνητό τους. Αυτό είναι ο βασικός στόχος, να μειωθεί η γραφειοκρατία και όλος αυτός ο φόρτος όσο γίνεται να περιοριστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει και τη μείωση του διοικητικού κόστους περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο κατανοητό αν δει ο καθένας τι ισχύει στην ε, κάθε χώρα. τεμποδίων κούρσα από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να μπορέσει να ταξινομηθεί ένα όχημα που υπάρχει ήδη σε κάποια άλλη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα, για ένα ήδη ταξινομημένο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ταξινόμηση σε μία χώρα να ισχύει για όλες. Αν ισχύσει αυτή η αρχή, τότε θα έχουμε ε, πετύχει μία μεγάλη νίκη. Και επίσης, τρίτος στόχος, ε, να ε, καταπολεμηθεί η κατάχρηση και η ε, κλοπή των αυτοκινήτων ή των στοιχείων τους εδώ είναι μια μεγάλη ε, κλιματική δραστηριότητα. Υπάρχει δυνατότητα στο άρθρο 5 υπό περιορισμένες συνθήκες, ορισμένες μάλλον συνθήκες, να ε, απορριφθεί η ταξινόμηση ή να μπορεί ένα κράτος μέλος να αρνηθεί και στην αιτιολογική σκέψη 6 όλα αυτά τα εξηγούμε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει την έννοια της συνήθους κατοικίας της λεγόμενης. Δηλαδή ξεκαθαρίζεται εδώ ε, ρητά και σαφώς που διαμένει ένας πολίτης και που έχει ταξινομηθεί ένα όχημα και που θα πρέπει να δοθεί η άδεια κυκλοφορίας. Είναι συγκεκριμένος ο ορισμός και ορίζεται καλά τι είναι η έννοια της συνήθους κατοικίας. Στο άρθρο 3 το αναφέρει αυτό ο κανονισμός. Και επίσης από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταβάλλεται ε, ε, μια προσπάθεια να υπάρχει ενιαία προθεσμία ακριβώ στον τόπο της συνήθους κατοικίας, το κράτος αυτό, θα πρέπει ε, αυτή η νέα ε, άδεια να δίδεται εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Από χώρα σε χώρα διαφέρει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση και σίγουρα θα συζητηθεί η πιο μικρή ε, περίοδος ήταν στη Δανία που βρήκα, είναι 15 μέρες. Το Βέλγιο έχει αυτό το εξάμεινο ήδη που προτείνεται εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπόλοιπε χώρε ε, είναι κάπου ενδιάμεσα, από δύο εβδομάδες μέχρι έξι μήνες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε μια λογική προθεσμία, ούτε πολύ ε, μικρή αλλά ούτε και ε, άπειρη, για να μην υπάρχει έδαφος για καταχρήσει και προβλήματα. Αυτή η πρόταση είναι στο άρθρο 4 Άλλο θέμα τώρα. Ηλεκτρονική ανταλλαγή ε, πληροφοριών στο άρθρο 7 μεταξύ των διαφόρων κρατών. Γι' αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ηλεκτρονική ε, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρμοδίων αρχών ταξινόμησης, δεν μπορεί να επέλθει αυτή η απλούστευση. Θα πρέπει να δώσει τη συμφωνία του το κράτος. Υπάρχουν βεβαίως διάφορες ε, αρμοδιότητες οι οποίες ξεχωρίζονται ε, αλλά να υπάρχουν ε, εγγυήσει για τα πρότυπα και να υπάρχει αυτή η ηλεκτρονική δυνατότητα. Δεν υπάρχουν προβλήματα εδώ, μόνο πλέον εκτίματα μπορεί να φέρει αυτό. Υπονοείται και η αμοιβαία αναγνώριση των εγγράφων ταξινόμησης και των τεχνικών ε, διατάξεων. Ακόμα και αν είναι διαφορετικά τα όσα ισχύουν σε κάθε χώρα για τον τεχνικό έλεγχο και για την έγκριση και για την ταξινόμηση, η προϋπόθεση είναι αμοιβαία αναγνώριση. Και σε αυτό ε, στοχεύει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επίσης ε, γίνεται λόγος και για μια προσωρινή άδεια για ε, μεταφορά σε ένα άλλο κράτος μέλος. Το άρθρο 6 οριζόνται αυτά και αφορά κυρίως τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τα οποία αγοράζει κάποιος σε μια χώρα και πρέπει να τα μεταφέρει σε μια άλλη. Και στο άρθρο 8 γίνεται λόγος και για τις αντιπροσωπείες ε, αυτοκινήτων και για ε, τους εξουσιοδοτημένους εμπόρους. Όλα αυτά συνιστούν μια πρόταση πάρα πολύ πρακτική και εφαρμόσιμη. Δεν νομίζω ότι χωράει εδώ πολύ μεγάλη κριτική. Ε, απλουστεύει πάρα πολύ τα όσα ισχύουν και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, γενικά με τους στόχους. Εγώ τι έκανα στις προτάσεις μου. Δεν προτείνω τόσο πολύ διόρθωση του κειμένου, αλλά ενίσχυσή του σε κάποια στιγμή, όσο και διευκρίνηση σε μερικά άλλα, για να ε, ξεκαθαριστούν ορισμένα θέματα που θεωρούσα ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Ε, αυτά εισαγωγικά. Και να σας πω τώρα εγώ ε, τι προτείνω, τι καλωσορίζω και τι ενισχύω. Αυτές οι προσπάθειες να μειωθεί ε, η γραφειοκρατία και να μειωθεί και το γραφειοκρατικό κόστος. Δηλαδή ε, να υπάρξει μια διαδικασία πιο απλή αλλά και πιο οικονομική. Δεύτερον, Θυμάστε που είχε κάνει μια γνωμοδότηση ο Μπράιν Σίμψον για τις 20 μεγαλύτερες ανησυχίες των καταναλωτών και των πολιτών. Ε, και αυτό το έχω συμπεριλάβει στην τροπολογία μου υπαριθμών 1 και στην τροπολογία υπαριθμών 2 για τις 20 κύριες ανησυχίες των επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών. Στη συνέχεια, θα πρέπει να στρέψουμε το κέντρο βάρους και είμαι ακράδαντα σε αυτό στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην οδική ασφάλεια. Θα πρέπει βεβαίω αυτή να μην διακυβευθεί. Δεν έχει νόημα, πιστεύω τώρα, να αρχίσουμε να προτείνουμε ε, πάρα πολύ ε, λεπτομερείς ρυθμίσεις ή να ορθώνουμε νέους φραγμούς, γιατί από χώρα σε χώρα διαφέρει πάρα πολύ η κατάσταση. Θα πρέπει πραγματικά να περιοριστούμε σε αυτή την πρόταση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι πραγματικά, απλώς, ας πούμε, αν φέρουμε 200 τροπολογίες, τουλάχιστον οι 100 θα περιπλέξουν την κατάσταση αντί να την απλουστεύσουν. Και θα ήθελα πραγματικά να προειδοποιήσω και το και να παρακαλέσω και τους σκιώδεις εισηγητέ, αλλά και τους υπολείπους συναδέλφους να φροντίσουν τις τροπολογίες να προτείνουν απλούστευση προς ε, το συμφέρον των ενδιαφερομένων ε, πολιτών. Άλλο θέμα. Θέλουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε μία συνεκτική προσέγγιση με το πακέτο για την οδική ασφάλεια. Λογικό δεν είναι ε, για να υπάρχει αυτή η απλούστευση χωρίς να σημαίνει κάτι τέτοιο μείωση της ασφάλειας στους δρόμους. ειδική δική ασφάλεια ε, και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις σε όλες τις χώρες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Γιατί αν επιτρέψουμε να κυκλοφορεί ένα αυτοκίνητο ε, και σε άλλα κράτη-μέλη χωρίς ε, νέα διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να είναι υψηλά αυτά τα πρότυπα σε όλα τα κράτη. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για μένα είναι να υπάρξει μια διευκρίνηση και αυτό το λέω στην τροπολογία υπαριθμών 5 για το τι γίνεται με το νόμιμο κάτοχο των εγγράφων ταξινόμησης. Νομικά δεν είναι υποχρεωτικό αυτό να ε, αφορά τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ε, δηλαδή δεν πρέπει να ταυτίζεται ο νόμιμος κάτοχος με τον οδηγό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις leasing ας πούμε ή άλλες καταστάσεις που είναι άλλος ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων και άλλος ο οδηγός. Επίση, στην ανταλλαγή των δεδομένων θα πρέπει να τηρούνται κάποια πρότυπα και ευχαριστώ τον επόπτη ε, προσωπικών δεδομένων που έκανε συγκεκριμένες προτάσεις ε, και τις έχω συμπεριλάβει και στις τροπολογίες μου. Τελευταίο. Σε ό,τι αφορά τις άδειες για τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων για τους εμπόρους, ε, θα πρέπει οι ε, εθνικές νομοθετικές διατάξεις να ισχύουν ε, και μόνο σε περίπτωση διασυνοριακής κυκλοφορίας να ρυθμίζεται χωριστά. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν την κυκλοφορία ε, στα κράτη-μέλη, αυτό είναι θέμα στο ιστορικό των κρατών μελών και κάποιες ειδικέ πινακίδες που έχουν τα αυτοκίνητα όταν ε, είναι στα χέρια των εμπόρων, αλλού είναι πράσινες, αλλού είναι γαλάζιες, εκεί δεν μπαίνουμε σε αυτά τα χωράφια, μόνο όταν υπάρχει διασυνοριακή κυκλοφορία. Ε, σας είπα, ε, για την προθεσμία, αν θα πρέπει να είναι έξι μήνες ή όχι. Εγώ το άφησα έτσι, δεν το αλλάζω το εξάμεινο που προτείνεται. Αλλά άμα θέλετε το συζητάμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Ένα ερώτημα τώρα που θέλω να απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά το άρθρο 5 ότι μπορεί να αρνηθεί μία ε, έγκριση, μία άδεια, ε, μία κρατική αρχή και πώς θα γίνει αυτό και πότε μπορεί να γίνεται όταν έχει παρέλθει η προθεσμία ελέγχου. Ωραία, το καταλαβαίνω. Και τι ε, συνέπεια θα έχει αυτό θα πρέπει να γυρίσει πίσω στη χώρα προέλευσης ο οδηγός με το αυτοκίνητο για να ξαναελεχθεί εκεί. Τι γίνεται όταν εκπνέει η προθεσμία και δεν έχει ρυθμιστεί. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή απλώς μπορεί να πάει σε ένα κέντρο ελέγχου στη χώρα που διαμένει, που δεν είναι η χώρα στην οποία έχει ταξινομηθεί το αυτοκίνητο, για να γίνει εκεί ο τεχνικός έλεγχος. Το χειρότερο και η πιο λάθος ε, ρύθμιση θα ήταν να γυρίσει στη χώρα προέλευσης βέβαια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλους τους Έχουμε ήδη συναντηθεί, έχω κάνει τα σχόλιά μου και προτείνω να είμαστε όσο γίνεται πιο ε, εύστοχοι στις προτάσεις μας και στις τροπολογίες να περιοριστούμε σε θέματα μεταφορών και όχι να γίνει ένα τεράστιο ευχολόγιο αυτή η υπόθεση των τροπολογιών. Δηλαδή νομίζω ότι όσο λιγότερα ζητούμε τόσο περισσότερο θα επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Πανιού. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κανονισμός αυτός που έχει να κάνει με την απλοποίηση της ε, εγγραφής των ε, οχημάτων με κινητήρα ανάμεσα στα κράτη-μέλη λαμβάνει υπόψη μια από τις πιο μεγάλες ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών όπως εκφράζεται ε, μέσα από την έκθεση της ΣΥΜΚΟ για τις 20 ανησυχίες, ε, ε, μάλλον σημαντικότερες ανησυχίες σε σχέση με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο θα μου επιτρέψετε να διαπιστώσω ότι το πρόβλημα της κνέου εγγραφής είναι ίσονο σημασίας η εγγραφή των οχημάτων που είναι βέβαια σύμμορφα δεν ε, παρουσιάζει πρόβλημα και η κοινοτική αποδοχή των ε, το γιοταχή και των οχημάτων είναι υποχρεωτική εδώ και χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο η νέα εγγραφή γίνεται άμεσα επί τη βάση ενός πιστοποιητικού ε, εγγραφής σύμμορφο προς την οδηγία 1999-37 ευρωπαϊκή κοινότητα. Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι αγαπητές συνάδελφοι η βιασύνη να είναι λογική εδώ για να βελτιώσουμε την ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει διάφορες νομοθετικές προτάσεις τον Απρίλιο με στόχο να πλαισιώσει καλύτερα τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με κινητήρα και των εμπορικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Ωστόσο και εδώ θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ο κανονισμός που σχετίζεται με την απλοποίηση τη καταγραφή των οχημάτων με κινητήρα ανάμεσα στα κράτη-μέλη άμεσα επηρεάζεται από αυτές τις νέες προτάσεις. Για παράδειγμα, η οδηγία που σχετίζεται με την περιοδικότητα των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων με κινητήρα θα υποχρεώσει διάφορες χώρε να αναθεωρήσουν τις νομοθεσίες του στον τομέα αυτό. Το να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε μηδέν αναγνώριση του τεχνικού ελέγχου Όπω το επιθυμεί ο κανονισμό μας, μέσα σε μια περίοδο βαθιάς, βαθιών αλλαγών σε διάφορες χώρες μέλη, δεν είναι πολύ λογική, στο βαθμό που το κλίμα εμπιστοσύνη που θα ήταν απαραίτητο για τη λήψη τέτοιων μέτρων απουσιάζει. Άρα λοιπόν προς χάρη συνοχή του συνόλου των διοικητικών μέτρων που προτείνονται εδώ, εγώ θα ήθελα αυτό το κείμενο να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν θα έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσει για το πακέτο του, των εθνικών ελέγχων, ε, όπως αυτό που τροποποιεί την οδηγία 1999 ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ε, καταγραφή των ε, οχημάτων και την πρόταση κανονισμού για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με κινητήρα και των σειρωμένων καθώς και της τοποποίησης σχετικής οδηγίας. Αυτή είναι η θέση μας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ντεμπάκερ. Στα αγγλικά. Θα ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πολύ καλή γνωμοδότηση για την Επιτροπή Μεταφορών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε πρωτίστως με τα θέματα των μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προσέφερε μια βιώσιμη πρόταση, ένα καλό εφαλτήριο, το οποίο ήταν και απολύτως απαραίτητο, διότι οι πολίτες νιώθουν την έλλειψη των διαφανών κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα είναι απαραίτητη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πάλι συγχαίρω τον εισηγητή, διότι ε, ασχολήθηκε με διάφορα ζητήματα που τράβηξαν και το δικό μας το ενδιαφέρον. Ε, θα πρέπει να συνδέσουμε αυτό το θέμα με το συνολικό πακέτο των οδικών μεταφορών. Ναι, επίσης, να δούμε τα πιστοποιητικά επαγγελματικών μητρών και τη διάρκεια των τριών μηνών. Καλή πρόταση και αυτή και σε σχέση με την αποτίμηση αντί για τέσσερα-δύο χρόνια. Ε, αναρωτιέμαι αν είναι εφικτά αυτά και ίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επεκταθεί για τι προθέσει τη αυτέ είναι οι παρατηρήσεις μου και τη ομάδα μου. Επίση, το ζήτημα προστασία δεδομένων για του φιλελευθέρου είναι ύψη σημασία, και πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε μια σχετική διάταξη και σε αυτή την πρόταση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ε, τη βαρύτητα της διοικητικής απλούστευσης, ε, της μείωσης της γραφειοκρατίας. Ακόμη και στο Κοινοβούλιο είναι να περιπλέκουμε απλά πράγματα. Λοιπόν, ε, τις διατυπώσεις πρέπει να τις μειώσουμε όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τις επιχειρήσεις, όπως σωστά μας είπε και ο εισηγητής. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να ελέγξει αν οι αρχές έκδοσης αδειών κυκλοφορίας εργάζονται βάσει αυτού του κανονισμού, διότι για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια για την επαναταξινόμηση, ούτως ή άλλως θα προκύψει καλύψουν το, τα ζητήματα και το θέμα τεχνικού ελέγχου είναι καθαρά εθνικό θέμα και άρα είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν την υπηρεσία με αποτελεσματικό τρόπο και πάλι με στόχο τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθου. Θα λάβουμε υπόψη τη σημερινή συζήτηση για την επεξεργασία των θέσεων μα και θα συνεχίσουμε τις συσκέψεις με τον εισηγητή ε, και του σχεδόν εισηγητές. Ευχαριστούμε κυρία Λίχτεμπεργκ. Ευχαριστώ. Εγώ χαίρομαι πάντα όταν έρχεται μια πρόταση για απλοποίηση στην Ευρώπη, ας πούμε για ε, δραστηριότητες ή σπουδές ε, είναι πιο εύκολες. Αλλά θα ήθελα από την αρχή να πω το εξή να το σκεφτούμε και να κοιτάξουμε πάρα πολύ πώς θα το εφαρμόσουν αυτό τα κράτη-μέλη. Διότι το έχουμε ξαναζήσει σε ε, απλουστευτικές διατάξεις, έρχονται τα κράτη-μέλη μετά και τα εφαρμόζουν κατά το δοκούν και τελικά δεν βγαίνει τίποτα λογικό και χρήσιμο για τον πολίτη. Θα πρέπει να το πούμε αυτό και να το τονίσουμε. Δεύτερον, ευχαριστώ τον συνάδελφο Πίρκερ που το, μιλάει και για το κταίο, εν πάση περιπτώσει για τα κέντρα τεχνικού ελέγχου ε, οχημάτων ότι παραμένει αυτό το παραθυράκι και θα πρέπει να κλείσει. Γιατί τι θα γίνει εάν απορριφθεί η ταξινόμηση. Τι θα γίνει, θα εξακολουθεί να έχει το παλιό, ε, την παλιά πινακίδα το αυτοκίνητο. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Ε, αυτό με το θέμα της, με τη συνήθη κατοικία θα ξαναβρούμε μπροστά μας το παλιό πρόβλημα που είχαμε με την Ιταλία. Ε, πέμπτη, δέκατη φορά το ζήσα τώρα πρόσφατα στη Νομική Επιτροπή, γιατί έχουν άλλο ορισμό στην Ιταλία για το συνήθι τόπο κατοικία ε, και δεν υπάρχει δυνατότητα μετά μεταφορά σε άλλο κράτο μέλο. Και συμφωνώ από το συνάδελφο, με τον συνάδελφο συγγνώμη, από τη Γαλλία, οπωσδήποτε σε κάθε ε, πλευρά να δούμε ε, το κατά πόσο αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να κυκλοφορεί, είναι κατάλληλο για την κυκλοφορία στους δρόμους. γιατί υπάρχει μια καχυποψία ε, πώς να το κάνουμε ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη, εάν ελέγχουν όλα με τον τρόπο που θα όφυλαν. Κάτι που μου λείπει λίγο από την πρόταση και δεν ξέρω αν μπορεί να μας το απαντήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αυτές οι ιστορίες έχουν πολλές φορές επιπτώσεις στις ασφάλειες των αυτοκινήτων, κυρίως όταν πρόκειται για τροχαία ατυχήματα. Ε, το έχετε σκεφτεί αυτό ε, και πώς θα το πείσετε για τους ελέγχους ή όταν λείπουν κάποια έγγραφα, όταν χρειάζονται διασταυρώσεις, πώς θα λυθεί αυτό με τις ασφαλιστικές εταιρείε. Και ένα τελευταίο, δεν πιστεύω ότι πρέπει να έρθουμε ε, τώρα, να, πιστεύουμε ότι θα κατακλειστούμε από ένα κύμα αιτήσεων για αλλαγή πινακίδας ή για μεταφορά. Οι φοιτητέ που σπουδάζουν σε ένα πανεπιστήμιο ε, εξωτερικού ε, δεν αλλάζουν πινακίδα, κρατάνε την παλιά, γιατί ας πούμε σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις στάθμευσης δεν τις πληρώνουν ποτέ και τις κλήσεις, γιατί ε, ξέρουν ότι δεν θα τους βρουν. Για να μην μιλήσω και για τις ευρωπαϊκές ε, πινακίδες άλλων χωρών που κυκλοφορούν στις Βρυξέλλες, γιατί και εδώ συμβαίνει και το έχω ακούσει πάρα πολύ. Αλλά για αυτοί, αυτοί που θέλουν να το κάνουν, να έχουν σαφείς κανόνες και ε, να ξέρουμε τι ισχύει και αν τα υποστηρίζει όλα αυτά και ο επόπτης προσωπικών δεδομένων, καλώς. Θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Βαντάλεν από την Επιτροπή των Περιφοριών, θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα φοιτητών που έχουν έρθει εδώ από το Ινστιτούτο Δημόσια Διοίκησης ε, του Πανεπιστημίου του Λάιντεν. Ε, καλωσορίσατε. Πίτερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Για μας το σημαντικότερο είναι να λειτουργεί η εσωτερική αγορά απρόσκοπτα, ε, να είναι πιο κοντά στον πολίτη. Πραγματικά είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση και υποστηρίζουμε πολύ τον εισηγητή ομάδα μας των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Είμαι περίεργος να ακούσω την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποιες τροπολογίες. Για ορισμένα άρθρα, ας πούμε, Έχουμε πρόβλημα με τη διερμηνία. Όχι. Έχουμε ένα ήχο που είναι πολύ ενοχλητικός, λέει η κυρία Λιχτεμπέργκερ, και ε, μεγαλώνει ένταση συνεχώς, δεν ξέρω. Είναι στη γερμανική διερμηνία αυτό. Και τα γαλλικά δεν έχουν καθόλου διερμηνία. <laughs> Εάν δεν έχουν Γάλλη διερμηνία να σταματήσω, δεν είναι δυνατόν. Ο πρόεδρος δεν ξέρω αν θα λυθεί αυτό γρήγορα. Τώρα είναι εντάξει. Τα γερμανικά είναι εντάξει τώρα. Γαλλικά. Γαλλική καμπίνα είστε μαζί μας. Uh, One of the booths has captured the French booth, apparently. Ποια άλλη καμπίνα κρατά ο Μύρου τη γαλλική. Μπορείτε να το ελέγξετε. Αυτό δεν... Αυτό είναι σαν διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, δεν είναι Παρίσι, καλησπέρα το Παρίσι. Okay, Peter, can we try again now, please? And what's this noise? Am I speaking too loud or no, no. Τώρα εγώ φταίω, λέει ο κύριος Μαντάντε, μιλούσα πολύ δυνατά. Όχι, όχι, αλλά είναι σαν να έχει ένα τριζόνι, ένα τζίτζικα με στα αυτή σου. Α, Καλά, εν πάση περιπτώσει. Ξαναρχίζω, Πρόεδρε, στα Ολλανδικά. όπω έλεγα προηγουμένω, για μα είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση, γιατί ε, διευρύνεται η ενιαία αγορά, εμβαθύνεται, έρχεται πιο κοντά στον πολίτη ε, και ε, φεύγουν όλοι οι φραγμοί και τα εμπόδια. Εμεί λοιπόν υποστηρίζουμε τον εισηγητή στην προσέγγιση του. Έχουμε όμω συγκεκριμένε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τι τροπολογίε και ιδιαίτερα αυτέ του εισηγητού για το ε, νέο κανονισμό. Ιδιαίτερα το 7 ε, για τους εμπόρους. Αυτή η περίοδος που προτείνει ο εισηγητής είναι το πολύ τρεις μήνες. Αλλά επειδή η αγορά έχει νεκρώσει ουσιαστικά, δεν αγοράζει κανείς καινούργια αυτοκίνητα και έχει μειωθεί πολύ και το εμπόριο στα μεταχειρισμένα. Και ε, κατά την άποψή μας θεωρούμε αυτό το τρίμηνο πάρα πολύ σφιχτή ε, προθεσμία. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ε, γίνεται με τις προτάσεις αυτές του εισηγητού και πώς αντιδράτε στην τροπολογία 7. Αυτό είναι σκόπιμο να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή ή δυσκολεύει τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριο Σκόχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Πίρκερ. Το πρόβλημά μου ήδη ακούστηκε. Έχει να κάνει με ένα πρόβλημα συνοχής που μπορούμε να έχουμε με την οδηγία για το κταίο, για το τεχνικό έλεγχο. Γιατί όταν αλλάζει ο ιδιοκτήτης και όταν ε, αλλάζει και η χώρα, ε, θα πρέπει να γίνονται ξανά τεχνικοί έλεγχοι. Δεν ξέρω, πρέπει να συνοηθούμε και πάλι με αυτό κύριε Πίρκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από, την Κομισιόν έχουμε τον κύριο Βόκερ. Καλώς ήρθατε στις μεταφορές, κύριε Βόκερ. Κανονικά είμαστε φιλικοί προς τους ανθρώπους της Κομισιόν, ειδικά μα δεν είναι από την DG Move. Σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε σε αυτήν την συνεδρία της Επιτροπής. Καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεσης, είναι πολύ θετικό νομίζουμε και εκτιμούμε αυτή την θετική προσέγγιση στην πρόταση της ε, Κομισιόν. Κατάλαβα ότι υπάρχουν ε, διάφορες τροπολογίες που στόχο έχουν να τελειοποιήσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν τις προτάσεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τις συζητήσουμε και περισσότερες δεν μας δημιουργούν πρόβλημα. Ερωτήσεις που ετέθησαν ε, τώρα αφορούν την, ε, επαγγελματική, την ισχύ μάλλον της επαγγελματικής γραφής της τριμηνιάς. Εμείς στο σχέδιο προτείνουμε να μείνει στην κατεξουδότηση πράξη. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει στο ποιο θα ήταν το κατάλληλο, λότερο μάλλον χρονικό διάστημα. Το άλλο θέμα που αφορά την περίοδο αναφοράς, εμείς προτείνουμε τέσσερα χρόνια και προτείνεται εδώ τα δύο χρόνια, αλλά πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο θα είναι πολύ σύντομο. Όπως ε, ήδη υπόθηκε, δεν είναι εφικτό να το συντάξουμε αυτό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλες ερωτήσεις. Δεν είμαι βέβαιος. Α, για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η πρόταση αυτή δεν αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω το θέμα των ασφαλίσεων σήμερα. Πάντως εν γέννη Είμαστε ευτυχείς που αναφέρθηκαν αυτά τα σημεία στη συζήτηση τη σημερινή και ελπίζουμε πως όλες οι αμφιβολίες θα ληφθούν αργότερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίρκερ, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Θέλω να ευχαριστήσω μόνο τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης κατά κύριο λόγο. Θα πρέπει να περιμένουμε το πακέτο για την ασφάλεια στις μεταφορές, τις αντίστοιχες διατάξεις και τις εφαρμοστικές για να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο και θα πρότεινα Βεβαίως να τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά, να τα έχουμε υπόψη μας και να τα αναμένουμε. Σε περίπτωση που αυτές οι διατάξεις έρθουν πανευρωπαϊκά, ε, εντάξει, θα πρέπει να περιμένουμε την εφαρμογή τους και την τήρησή τους, σίγουρα. Μπορεί κανεί να διαφωνεί και θα πρέπει να το καθυστερήσουμε τόσο πολύ μέχρι να εφαρμοστούν, μέχρι να ελεγχθούν όλα αυτά και να τεθούν σε ισχύ και αν ισχύουν και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη και μετά να αντιδράσουμε. Όχι, εγώ προτείνω ε, να δείξουμε εκ των προτέρων μια θετική στάση και μια εμπιστοσύνη για να πούμε ότι εντάξει, όταν έρθουν όλες οι διατάξεις και εφαρμοστούν, καλώς. Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς είναι να απλοποιήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα την κατάσταση και διοικητικά και οικονομικά είναι ελάφρυνση για τους πολίτες. Ε, χωρίς ε, να απεμπολίσουμε ή να χάσουμε το θέμα της οδικής ασφάλειας. Ε, θα κάνουμε συζητήσεις και περιμένω και τις προτάσεις σας για τροπολογίες. Αλλιώς σας ευχαριστώ για τη συμφωνία που υπάρχει και τη συναντήληψη σε μεγάλο βαθμό σε όλο το φάσμα των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ. Κύριε Βαντάλεν, τι έχετε διαδικαστικό. Ναι, Πρόεδρε. Δεν θέλω να δυσκολέψω τη ζωή στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν είναι και από τη Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ αλλά εγώ ρώτησα κάτι για την τροπολογία 7 του εισηγητού ε, για τους εμπόρους και την απόδειξη που πρέπει να δώσω. Δεν ξέρω, μήπως δεν είναι η δική σας ε, τώρα υπόθεση να μου απαντήσετε, αλλά γραπτός ή να το διαβάσετε αρμοδίως, σας παρακαλώ. Κύριε Κόρκο, μπορείτε να απαντήσετε αυτό σήμερα ή γραπτός. Λοιπόν, σύντομα ανέφερα το σημείο αυτό, ότι δηλαδή η πρόταση της Επιτροπής ως έχει προτείνει να παραμείνει αυτό στις κατοξιδότητες συμπράξεις και ότι δεν έχουμε καταλήξει στη διάρκεια, για τη διάρκεια της ε, εγγραφής των επαγγελματικών οχημάτων. Θα πρέπει να το μελετήσουμε να δούμε ποια περίοδος θα είναι η καταλληλότερη. Μάλιστα. Το σκέφτονται ακόμα δηλαδή. Ωραία συνάδελφοι. Λοιπόν, η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 16 Οκτωβρίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών προβλέπεται για τις 27 ε, Νοεμβρίου. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η ημερομηνία της ψηφοφορίας στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, αλλά η ημερομηνία κλειδί είναι 16 Οκτωβρίου καταρχήν, ως προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Ευχαριστώ και περνάμε στην επόμενη έκθεση που είναι το πακέτο των ρολιμένων και των χρονοθυρίδων. Έχουμε ένα κομμάτι αυτού του πακέτου λοιπόν και ο εισηγητής είναι ο κ. Ουτζίας που έχει και το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Σίμψον. Σας ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις πολυάριθμες τροπολογίες που υπέβαλαν. Ε, είναι πάνω από 300. Και αυτό επιβεβαιώνει την μεγάλη σημασία που αποδίδουν όλες οι πολιτικές ομάδες στο θέμα των ε, χρονοθυρίδων. Βέβαια, για λόγους χρόνου δεν θα μπορέσω να μπω στην ουσία κάθε μιας ε, τροπολογίας που έχει υποβληθεί. Και ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους, όμως θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι έτοιμοι για πιθανή ε, να, για υπεραιτέρω εξηγήσει ε, μέσα στη συνεδρίαση των ε, σκιωδών, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων, είτε μέσω διμερών επαφών. Θα πρέπει να, επίσης να σημειώσουμε πώς οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν αγγίζουν σημεία ευαίσθητα του θέματος λόγω της αύξησης του ορίου χρήσης στο 85% ε, προς 15% αύξηση της σειράς ε, που περνά από την ε, τιμή κράτησης της χρονοθυρίδας. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζονται τα θέματα των ε, δεσμεύσεων των αερολιμενικών αρχών που στην ουσία ε, επαναφέρουν το status quo. Εγώ πιστεύω πως ε, θα πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για να φτάσουμε μια υψηλού επίπεδου συμβιβαστική λύση που θα μπορεί να δώσει μια πραγματική βελτίωση των, της χωρητικότητας των αερολιμάνων και ε, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ε, της βιομηχανίας, της αεροναυτιλίας. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι με μεγάλο συνέστημα ευθύνη ε, να, να πιέσουμε την Κομισιόν για να δώσει ανταπόκριση στα απαιτήσει τις οποίες υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό και θέλω να στηρίξω τη δράση της Κομισιόν σε αναζήτηση μιας συμβιβαστική εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και με το Συμβούλιο για τις πτυχές που είναι πιο σημαντικές για αυτό το θέμα, δηλαδή το μάκρος των σειρών και την αύξηση του κατοφλίου χρήσης των χρονοθυρίδων. Να πω αμέσως ότι στόχος μου είναι να ενημερώσω τους συναδέλφους πως έχω φτιάξει έναν οδικό χάρτη προσέγγισης στην ψηφοφορία της Επιτροπής που προβλέπεται στις 6 Νοεμβρίου και ότι θα προχωρήσουμε μέσω της σύγκλησης δύο τεχνικών ε, τραπεζιών συζήτησης ε, με, βάση αυτή την, ε, με αρχή αυτή την εβδομάδα και μια συνεδρίαση των σκεωδών που προβλέπεται για τις 26 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο σύμφωνα με τις δεσμεύσεις ε, που έχουν ήδη εκδηλώσει οι συνάδελφοι. Θέλω αμέσως ε, να μιλήσω για το θέμα της, ε, του μάκρους των σειρών των χρονοθερίδων. Όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν υποβάλει τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν. Όσον αφορά το όριο χρήσης των χρονοθερίδων, μείωση από 15 σε, την καλοκαιρινή περίοδο σε 10 το χειμερινή περίοδο και σε 5 μάλιστα και με βάση τις τοπικές συνθήκες που επιτρέπουν την μείωση ή την αύξηση της σειράς σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε ρολιμένα. Πολλές τροπολογίες θέλουν δεν να ακυρώσουν τη διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στην καλοκαιρινή περίοδο και την χειμερινή περίοδο, ζητώντας οι σειρές να μείνουν πέντε, όπως προβλεπόταν από τον προηγούμενο κανονισμό. Φαίνεται δε ε, να επιβεβαιώνεται η διατήρηση του δεσμού της συνέχισης ε, μιας σειράς χρονοθυρίδων για να παραμείνει μέσα στο πνεύμα των κεκτημένων δικαιωμάτων που θα πρέπει να πετούν στις πέντε θηρίδες που έχουν προβλεφθεί, διαφορετικά κινδυνεύουν να τις χάσουν. Ε, κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο να βρούμε μια συμβιβαστική για αυτό το σημείο όλες οι ομάδες συμφωνούν στο να προσφύγουμε στους τοπικούς ε, κανόνες με βάση, ε, μάλλον όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποπτία των ε, χρονοθυρίδων, αλλά έχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την χρήση των σειρών. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι υπάρχει σχεδόν ομόφωνη γνώμη όσον αφορά του Network Airport, που είναι ένας οργανισμός που θέλει να περάσει μη δεσμευτικούς, ε, μη, μη δεσμευτικούς κανόνες για την διαβίβαση στοιχείων των αεροπορικών εταιριών, πράγμα το οποίο μπορεί κάλλιστα να κάνει ο Ευρωκοντρόλο, υπάρχουν οργανισμός. Όσον αφορά τους όρους ε, για τον συντονισμό των αεροδρομίων, βασικός στόχος είναι να αποδυναμωθούν οι διατάξεις της Κομισιόν για τον καθορισμό ενός ε, συντονισμένου αεροδρομίου. Ιδιαίτερα οι συνάδελφοι του ΕΛΚ, οι συντηρητικοί και διάφορες ε, τροπολογίες έχει υποβάλει η κυρία Φώστερ, ζητούν ενίσχυση του ρόλου της Κομισιόν ως διαχειριστή του δικτύου και έτσι να περιορίζεται η θέση της όσον αφορά τον καθορισμό του, του συντονισμένου αεροδρομίου. Ωστόσο δεν νομίζω πως υπάρχει εδώ ακόμα συμβιβαστική λύση. Μετά από την συνάντηση δε των συντονιστών, ένα σημείο το οποίο αποκτά μεγάλη σημασία είναι η ανάγκη να εγγυηθούμε ότι η δραστηριότητα των συντονιστών θα χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαφάνεια. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο βρήκε σύμφωνος ε, όλους τους συναδέλφους και ε, για το συγκεκριμένο θέμα. Η πρόταση αυτή αφορά μεγαλύτερη ανεξαρτησία των συντονιστών, όπως και εγώ είχα εκφράσει την επιθυμία στο σχέδιο έκθεσης, κυρίως μέσω διαδικασιών πιο διαφανών όσον αφορά τη διαχείριση των στοιχείων συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών, που προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμες υπό τη μορφή ατομικών στοιχείων και όχι μόνο ομαδοποιημένων, όπως προβλέπεται από την Κομισιόν αρχικά στην πρότασή της. Επίσης, χαίρομαι για το γεγονός ότι ως προς αυτό διάφοροι συνάδελφοι Ματσίκεβιτ, Ζαζάντα, Μαρινέσκο, Τικάου και Ρίκε έχουν επιβεβαιώσει μέσω των τροπολογιών τους την έννοια της ε, οικονομικής σχέσης που ο συντονιστής πρέπει να υποβάλει για κάθε περίοδο κυκλοφορίας έτσι ώστε να μπορούν τα μέρη που συμφωνούν για τη χρηματοδότηση, δηλαδή αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες, να έχουν πλήρη πρόσβαση στη δραστηριότητα των συντονιστών με σε μια οπτική μέγιστης διαφάνειας. Το πέμπτο θέμα είναι αυτό που αφορεί αφορά τον κανόνα 80 προς 20. Η πρόταση της Κομισιόν, όπως επιβεβαιώνεται στον Τουσιέ, να αυξηθεί δηλαδή το κατόφλι χρήση των σλότ από το 80% στο 85% αποτέλεσε αντικείμενο ανησυχητικών επικρίσεων από όλε τις ομάδες που υπέβαλαν τροπολογίες που στόχο έχουν να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς του 80 προς 20. Από την εξέταση των τροπολογιών που υποβλήθηκαν ωστόσο δεν προκύπτει μια πιθανή λύση εναλλακτική. Και αυτό το λέω γιατί οι συνάδελφοι χωρίς να, να ξέρουν ότι αν δεν ανατρέξουμε σε μεγαλύτερη χρήση των ε, εδαφών θα επιτρέπει να αυξηθεί η χωρητικότητα των ευρωπαϊκών αερολιμένων. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως η πρόταση της Κομισιόν, εάν εγκριθεί, θα εγγυόταν μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση στα κορεσμένα, ε, των χρονοθυρίδων στα κορεσμένα αεροδρόμια. Όλοι οι συνάδελφοι τώρα του ΕΛΚ παρατάσσονται κατά της κράτησης των χρονοθυρίδων που θεωρούν ότι είναι πολύ δαπανηρή για τις αεροπορικές ιστορίες. Ενώ ορισμένοι σοσιαλιστές συνάδελφοι, για παράδειγμα, στην, έκθεση, στην τροπολογία 244 του κυρίου Σασόλ, είναι υπέρ των κυρώσεων για εκείνους τους φορείς που καθυστερημένα επιστρέφουν τις χρονοθυρίδες. Νομίζω πως η υιοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου, όπως βλέπουμε από την αξιολόγηση αντικτύπου που έχει κάνει η Κομισιόν, θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για να αποθαρρυνθεί η η χαμηλή χρήση των, ή μάλλον η κατάλληλη χρήση των σλότ, αλλά θα πρέπει να επικυρωθεί. Η περαιτέρω δε ε, Επίσης θα πρεπει να επικυρωθει η δε επισης θα καταστησει πιο αυστηρούς τους κανόνες του άρθρου 18 που αφορά τις κυρώσεις. Ακόμα ένα σημαντικό θέμα είναι ο νομικός καθορισμός των χρονοθυρίδων που εμείς οι ευρωβουλευτές ε, θα πρέπει να ασκήσουμε πλήρως το νομοθετικό μας έργο και να εισάγουμε το, νομοθετικό ορισμό της χρονοθυρίδας που θα συνοδεύσει τη τεχνική και επιχειρησιακή περιγραφή που περιλαμβάνεται ήδη στους προηγούμενους κανονισμούς. Γνωρίζω πως υπάρχουν ε, δράσεις συντηρητικές και ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι θα ήθελαν να μην αντιμετωπίσουν τη δυσκολία που σημαίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ωστόσο πως είναι δυνατόν με μια σειρά συμβιβαστικών να βρούμε έναν ορισμό ώστε να καταφέρουμε να βρούμε δηλαδή μια διατύπωση που να μπορέσει να βρει σύμφωνους όλους όσους θέλουν να δεχτούν αυτή την πρόκληση. Να τονίσω επίσης τη θετική ε, συμβολή της συναδέλφου Εύα Λίχτεμπεργκ με την τροπολογία 201 στην ουσία επιβεβαιώνει την ανάγκη ύπαρξης ε, και της ε, χρονοθυρίδας ζητώντας να συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι νομικοί αρμόδιοι. Τελευταίο σημείο αφορά την μεταφορά και την ανταλλαγή των χρονοθυρίδων. Όσον αφορά τη δευτερογενή αγορά, από πλευρά ορισμένων συναδέλφων Γάλλων, Βιράκ και Ταντέν με την τροπολογία 250, η πλειοψηφία φαίνεται να επιβεώνει αυτή την πράξη που ήδη χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες εδώ και χρόνια. Βεβαίω, η ανταλλαγή χρονοθυρίδων μέσω οικονομικού αντισταθμίσματος θα πρέπει να γίνεται μέσω ε, κανόνων που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια. Και εδώ είναι σκόπιμες οι τροπολογίες 262 και 269 που υπέβαλαν οι συνάδελφοι Φιντάντζα και Καντσάν που στόχο έχουν να εμποδίσουν τις εταιρείες να μεταφέρουν ε, χρονοθερίδες με κερδοσκοπικό σκοπό αμέσως μετά από την χορήγησή τους και αφού και πριν καν να την έχουν χρησιμοποιήσει τη χρονοθερίδα τους. Άλλες τροπολογίες όπως οι 270 Σασόλη, 271 Φιντάντσα Καντσάν και η τροπολογία Σερακιάν στόχο έχουν να ε, χρησιμοποιηθούν τα πρόσοδα του, της πώλησης των χρονοθυρίδων στην βελτίωση των υποδομών, όπως προτείνεται και στο σχέδιο έκθεσης. Οι συνάδελφοι προτείνουν πως αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο διαχείρισης από την ανεξάρτητη αρχή που προβλέπεται από την Οδηγία 12-2009, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω διοικητικός φόρτος. Και αυτή η πρόταση πιστεύω πως είναι λογική. Τέλος, Πρόεδρε Σίμψον, σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Νομίζω πως υπάρχουν όλες οι προποθέσεις για να βρεθεί μια καλή συμβαστική λύση με τους συναδέλφους που συνεισέφεραν με τις απόψεις τους σε αυτή την πρώτη φάση. Σας ευχαριστώ κύριο Τζίος, ο κύριος Φιντάντζα από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε πάνω σε αυτό το δύσκολο θέμα. Έδωσε μια εικόνα πολύ σωστή για τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν και για τα πιο σημαντικά σημεία. Έχουμε ήδη κάνει συζήτηση σε αυτά τα βασικά θέματα επανειλημμένως. Εγώ θέλω απλά να επαναλάβω κάποιες θέσεις που απαντήθηκαν και μέσω των τροπολογιών που υπέβαλαν οι συνάδελφοι της ομάδας του ΕΛΚ. Όσον αφορά τον κανόνα του χρησιμοποίησε το ή χάσε το. Ε, από την ομάδα μας ε, είναι αρνητική η γνωμοδότηση όσον αφορά την πρόταση τροποποίησης της Κομισιόν γιατί θεωρούμε πως το πέρασμα από το 80 ε, προς 20 στο 85 προς 15 δεν λύνει το πρόβλημα της αύξησης χωρητικότητας, πρόβλημα το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Είναι ένας δρόμος που τεχνικά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και επίσης όπως γνωρίζουμε θα οδηγούσε σε μια έλλειψη ισορροπίας ε, γενικά ανάμεσα στους κανόνες δηλαδή που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και τους κανόνες που ισχύουν στον υπόλοιπο κόσμο. Πιθανότατα θα είναι απαραίτητη μια περαιτέρω προσπάθεια, όχι μόνο από το Κοινοβούλιο και συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, προσπάθεια και από πλευράς της Κομισιόν για να αναζητήσουμε άλλους τρόπους αύξησης τη ε, αερολιμενικής χωρητικότητας όσον αφορά το μάκρο των σειρών, των χρονο και από πλευρά μα φάνηκε μια βούληση μάλλον διάχυτη να διατηρηθεί μια πρόβλεψη πέντε εβδομάδων. Εγώ θα άφηνα στην συμβιβαστική φάση το θέμα τη ε, συνέχεια, τη διαδοχικότητα. Έπειτα υπάρχει και αρκετά ευρεία συμφωνία όσον αφορά την ανάγκη αξιοποίηση τη χρήση των τοπικών κανόνων, local rules, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένε και πολύ καλά καθορισμένε περιπτώσει, Αλλά να αφήσουμε μια κάποια ευελιξία αξία Εδώ θα είναι χρήσιμο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα αεροδρόμια που αντικειμενικά βρίσκονται σε κατάσταση κορεσμού ή πολύ έντονη συμφόρηση. για τη χρηματοδότηση των συντονιστών. Και εγώ έχω κάνει εδώ μια διαβούλευση ανάμεσα στις τροπολογίες των διαφόρων πολιτικών ομάδων που στόχο έχουν να εγγυηθούν μεγαλύτερη διαφάνεια για την χρηματοδότηση είναι σαφέ ότι με βάση τη σημερινή κατάσταση είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι μια τρίτη ε, μονάδα ή οντότητα θα μπορεί να εγγυηθεί την πληρωμή και την πληρωμή του συντονιστή. Πρέπει δηλαδή να βρούμε μια κατάσταση όπου οι εταιρείε και οι αερολιμένες ήταν όλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβάλλουν για να πληρώνεται ο συντονιστή. Ίσως θα μπορούσαμε να δουλέψουμε ώστε οι μηχανισμοί αυτοί να γίνονται πιο διαφανείς, να καταστούν πιο διαφανείς και να εγγυηθούμε και μεγαλύτερη ανεξαρτησία για τον συντονιστή. Να επαναλάβω και το ανέφερε και ο κύριος Ούτζας ε, ότι ε, ακούστηκαν επικρίσεις όσον αφορά το τέλος κράτησης της χρονοθυρίδας. Εμείς είμαστε υπέρ του να τιμωρούνται οι κακές συμπεριφορές μέσω ε, κυρώσεων πιο συγκεκριμένων και πιο αποτελεσματικών. Le compagnie aeree con una tassa di prenotazione έτσι ώστε να είτε είναι εταιρείε οι οποίε σωστά χρησιμοποιούν τι χρονοθυρίδε του, είτε είναι εκείνε που κακά χρησιμοποιούν τι χρονοθυρίδε του, να μπορούν να επιβληθούν κάποιε κυρώσει. Είμαστε υπέρ δηλαδή των πιο αυστηρών και πιο αποτελεσματικών κυρώσεων. Και όχι υπέρ του τέλου κράτηση τη χρονοθυρίδα. Τώρα, ο εισηγητής προτείνει μια διάμεση λύση μέσω τη βάση δεδομένων για πληροφορίες για κάποια αεροδρόμια και εδώ πιστεύω πως θα βρούμε μια συμβιβαστική λύση αλλά θεωρούμε πω είναι απαραίτητο να μην επιδεινωθούν, να μην επιβαρυνθούν από γραφειοκρατικά περισσότερο ε, τα αεροδρόμια και οι ορισμοί αυτών. Παραμένει ανοιχτό και στο εσωτερικό τη ομάδα μα το θέμα της του νομικού ορισμού των ε, ε Θα πρέπει να βρούμε έναν ε, ορισμό ώστε να μπορούμε να ορίσουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης κάθε χρονοθυρίδας. Η χρονοθυρίδα είναι ένα περίεργο αγαθό το οποίο έχει γίνει αντικείμενο εμπορίου ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν το έχουν καν στην κατοχή τους, δεν είναι οι κάτοχοι του δικαιώματος αυτού. Είναι δύσκολο λοιπόν να καταλάβουμε, αλλά θα το δούμε αυτό, κατά πόσο ο ορισμός που προτείνει ο εισηγητής θα είναι μια σωστή απάντηση. Τελευταία πτυχή και κλείνω Πρόεδρε όσον αφορά τη δευτερογενή αγορά, το second training, trading και από πλευρά των συναδέλφων δουλέψαμε ώστε να καταστεί πιο διαφανής η δευτερογενής αγορά. Στην ομάδα μας έχουμε μια θέση πολύ στεναρή από πλευρά των Γάλλων συναδέλφων, οι οποίοι θέλουν να κόψουν από τη ρίζα τη δυνατότητα ύπαρξης μιας τέτοιας δευτερογενούς αγοράς. Ε, στην ουσία το συζητάμε στην ομάδα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρχει η δευτερεύουσα αγορά, αλλά να είναι διαφανής, ρυθμισμένη. Και να μην επιτρέπει έτσι η δημιουργία μιας κερδοσκοπικής ε, χρηματοπιστωτικής αγοράς που δεν έχει καμία σχέση με την αύξηση της χωρητικότητας των αερολιμένων. Επ' αυτού λοιπόν θα κάνουμε προτάσεις ε, και θα είμαστε ανοιχτοί για συμβαστικές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σασόλη τώρα από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια στον κύριο Ούτζες. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και κυρίως να τον ευχαριστήσω γιατί δέχτηκε κάποιες από τις τροπολογίες που παρουσιάσαμε. Να μιλήσω καταρχήν για την ανεξαρτησία του συντονιστή. Φυσικά, όπως όλοι οι βουλευτές, στηρίζω την μέγιστη ανεξαρτησία του συντονιστή, τη μέγιστη διαφάνεια της ε, διαδικασίας ε, χορήγησης των χρονοθυρίδων είναι πολύ σημαντικό να εισαχθεί ένας κανόνας για την επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων και την αποφυγή αυτών για τους φορείς που ενδιαφέρονται λοιπόν για τη χορήγηση των χρονοθυρίδων. Και έχω υποβάλει σχετικές τροπολογίες. γεννής αγορά τώρα. Είμαι υπέρ αλλά με κανόνες που να εγγυώνται τη διαφάνεια και τη σαφήνεια. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να ένα κομμάτι των προσόδων της δευτερογενούς αγοράς να ε, να προορίζεται για την ε, τεχνολογική πρόοδο και για την ε, βελτίωση των υποδομών. Κάτι τέτοιο πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε αυτά να τα αναθέσουμε σε ένα ταμείο το οποίο θα διαχειρίζεται κάθε κράτος μέλος από, και μάλιστα η αρχή ρύθμισης των μεταφορών που προβλέπονται από την οδηγία 12 του 2009 και ως προς αυτή την κατεύθυνση έχω υποβάλει τροπολογίες. Το αεροδρόμιο τώρα ενσωματωμένο σε το δίκτυο. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία αεροδρομίων μάλλον να μην δημιουργηθεί νέα, νέα ε, κατηγορία αεροδρομίων γιατί μπορεί έτσι να περιπλακούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Τώρα, ο κανόνας 80 προ 20 και η σειρά των χρονοθυρίδων. Πρέπει να ξαναδούμε την πρόταση της Κομισιόν σε ορισμένα σημεία. Συμφωνώ για τον κανόνα 85-15 δεν είναι όλοι οι βουλευτές υπέρ της διατήρησης του κανόνα 80-20. Εμείς είμαστε υπέρ του κανόνα 85 προς 15, ενώ ταυτόχρονα ε, να συνδυάζεται με πιο μακρές σειρές διαδοχικές και μακριές ε, θα είναι αυτό εξαιρετικά δύσκολο και για τις εταιρείες που έχουν τις χρονοθυρίδες αλλά κυρίως για τις νεοεισερχόμενες εταιρείες. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Κατά γνώμη μου θα πρέπει να διατηρήσουμε τη σειρά των πέντε χρονοθυρίδων αλλά να εισάγουμε την διαδοχικότητα. Ε, εκεί όπου είχαμε δηλαδή περιόδους ιδιαίτερης συμφόρησης σε κάποιον αερολιμένα θα μπορούσαμε να επιμηκύνουμε τη σειρά των χρονοθυρίδων μέσω των local rules. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε διαχείριση της χωρητικότητας των αερολιμένων με αποτελεσματικότερο τρόπο και άρα καλύτερη χρήση των χρονοθυρίδων. Για τον κανόνα 85 προς 15 είδα από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν ότι πολλοί συνάδελφοι είναι υπέρ της διατήρησης του κατοφλίου 80 προς 20. Εγώ αντιθέτως πιστεύω πως μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση της Κομισιόν διατηρώντας ε, τη σειρά των πέντε χρονοθυρίδων αν είναι ε, διαδοχικές. Δεν θα υπάρξουν διαφορές στην ευελιξία που δίνονται, δίνεται στις ε, αεροπορικές εταιρείες, ενώ διαφορές θα υπήρχαν εάν υπήρχε ανάγκη επιμήκυνσης της σειράς των χρονοθυρίδων. Θα ήταν ωστόσο χρήσιμο κατά τη γνώμη μου και κλείνω έτσι και με μια οπτική διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και θα μπορούσαμε ίσως και να το κάνουμε αυτό όλοι μαζί, να βρούμε μια θέση κάπως πιο θεραλέα, ε, για ένα κείμενο πιο φιλόδοξο. Ευχαριστώ. Λίχτεμπεργκερ. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα θα πρέπει πάντα να έχουμε προοφθαλμού ότι πρόκειται για ένα πολύ μικρό ποσοστό των χρονοθυρίδων. Δεν είναι μια γενική νέα ρύθμιση του συστήματος χρονοθυρίδων. Ε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ε, και θα ήθελα να επανέλθω και να πω το εξή. Για μένα υπάρχουν μερικά σημεία που παρόλα αυτά ε, καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν. Το ένα είναι αυτό που το είδαμε την κρίση με το ηφαίστειο ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία διαχείριση και κράτηση των εισιτηρίων ε, τρένου και αεροπλάνου. Και ε, στην περίπτωση αυτή των χρονοθυρίδων, λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται και με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια. Γιατί δεν λαμβάνονται αρκετά υπόψη αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η αέρια κυκλοφορία. Και το θέμα της χρονοθυρίδα, τι εστί χρονοθυρίδα. Ακούσαμε ολόκληρη διάλεξη ε, ότι είναι ένα άειλο αγαθό της ανθρωπότητας ε, που κάποιος μας το δίνει, το μοιράζουμε, το πουλάμε, ξέρω εγώ. θα πρέπει να βρεθεί ένας ορισμός ε, που να ορίζει ότι είναι δημόσιο αγαθόν και η κατανομή θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια διαφανή και ε, σεβόμενα και το περιβάλλον. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμπάκερ. Eh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο θέματα που θέλω οπωσδήποτε να προσθέσω για να πω στον εισηγητή. Ε, είναι καλή δουλειά του αλλά δύσκολη ε, δύο σύντομα που θέλω να τονίσω. Πρώτον, θεωρώ σημαντικό να πούμε ότι η όλη συζήτηση που κάνουμε τώρα γίνεται και διεθνώς, έτσι, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Έχω την εντύπωση ότι εμείς ομφαλοσκοπούμε υπερβολικά, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν και διεθνείς επιπτώσεις. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους και στον εισηγητή να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, ε, πολύ. Ε, ιδιαίτερη ε, κλάδη της ε, αεροπλοείας είναι οι επιχειρηματίες που πετούν με δικά τους αεροσκάφη και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μικρά περιφερειακά αεροδρόμια αλλά και με μεγάλους αερολιμένες και έχει να κάνει και με την οικονομική ζωή. Τι γίνεται λοιπόν με την business aviation, με τις χρονοθυρίδες, αν υπάρχει μια συγκεκριμένη υποδομή, γιατί στο παρελθόν έχουν γίνει επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί και να είναι σε θέση να ασκεί τις κανονικές της δραστηριότητες και αυτή η εναερία κυκλοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την Επιτροπή, ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να χαιρετήσω τους παρισταμένους. Ε, ελπίζω να μην βασίζεστε στον πίνακα βαθμολογίας της Eurovision, γιατί εμείς θα παίρναμε σίγουρα μηδέν βαθμούς. Σας ευχαριστούμε κύριε Ουγγίας για την έκθεση καθώς και για τις τροπολογίες για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρονοθυρίδες. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά ο στόχος εδώ είναι να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή χρήση της χωρητικότητα των ρολιμένων μας. Αλλά είμαστε κατακαιρματιστές εισαγωγικά. Προσπαθούμε ε, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα χωρίς όμως να αυξηθεί και το κόστος. Αυτό είναι το modus operandi. Ε, τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης, πως από ό,τι φαίνεται γίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή Μεταφορών, από τα περισσότερα μέλη τουλάχιστον για τη δευτερογενή αγορά, για το θέμα της οξυμένης διαφάνειας, ε, και της ανεξαρτησίας των συντονιστών ε, της κατανομής ε, χρονοθερίδων. Δεν θέλουμε να είμαστε ριζοσπαστικοί, να μιλάμε για κατάσχεση χρονοθερίδων κτλ. Όλα αυτά δεν τα αγγίζουμε καν, γιατί έτσι αυτή είναι και η πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Όμως προκύπτει από τις τροπολογίες ότι υπάρχουν διάφορες ανησυχίες, διακομματικές θα έλεγα, σε σχέση με την πρότασή μας, που σχετίζονται με το 80-15 και την παράταση των σειρών χρονοθυρίδων. Αυτά τα δύο ζητήματα εξετάζονται από κοινού συνήθω ε, και νομίζω ότι ε, μέσω αυτών αφαιρόσασταν. Ε, καλό θα ήταν ενδεχομένω να διαχωρίσουμε αυτά τα ζητήματα τελικά για τι μακριέ σειρέ χρονοθυρίδων. Εξετάσαμε όλου του εναλλακτικού τρόπου και συγκεκριμένα τι σειρέ των 7 χρονοθυρίδων. Κάναμε αξιολόγηση αντικτύπου που δείχνει ότι δεν ήταν και πολύ σημαντικά τα ωφέλη θέλει. Α, κάποιοι αερολιμένες επιθυμούν να διατηρήσουν τις ε, μακριές σειρές 10-15 όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα δεν θέλω να καταθέσω συμβαστική πρόταση, όμως αν εξετάσουμε θεωρητικά το ζήτημα και αν διατηρήσουμε την σειρά των 5 και αυτός είναι ο γενικός κανόνας, ε, εν τη αυτή περιπτώσει, όπως ο κύριος Φινάνσα και ο κύριος Σακόλη μας είπαν, ε, θα συνηγορούσαμε υπέρ του να δοθεί μία ευκαιρία στους αερολιμένες για να εφαρμόσουν και τους τοπικούς κανόνες. Αλλά και πάλι να σας πω ότι αεροδρόμια όπω το η Λισαβόνα, Ντίσσελντορφ, ε, Παρίσι Αλντεγκόλ, της Ρώμης, το αεροδρόμιο της Ρήγης θα υποφελούνταν από την ε, νέα μέθοδο, αλλά άλλα αεροδρόμια πάλι όχι. Ε, βάσει τη δική μα πρόταση, αν παρατείνουμε τη σειρά, ε, ε, θα έχουμε τους ε, τοπικούς κανόνες σε 9 ερολιμένες, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε επιτύχει μόνο το ίμιση του στόχου μας, έξω και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν εδώ και κάποιοι προκρίνουν ως γενικό κανόνα να έχουμε συντομότερες σειρές, κάτω των 5. Σε σχέση, Πρόεδρε, με αυτά που είπατε για το 75 15 σε σχέση με την χρήση, ε, κατά τη διαστολή με το σημερινό 80-20 σε διάφορα φόρα είχαμε ε, επικρίσεις και είπαν ότι το 85-15 αντιβαίνει στις διεθνείς ε, πρακτικές ε, διότι τίθεται και το ζήτημα των τρίτων χωρών και επιτρέψτε με να αναφερθώ σε κάποια από τα επιχειρήματα αυτών που αντιτάσσονται στο 85-15. Τι σημαίνει σε συμφορημένους ρολιμένες αυτό σημαίνει ότι οι τρίτες χώρες με οποίες επικοινωνούν δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 80-20. Δηλαδή δεν υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα ε, στους Σε σχέση με την, κανόνε τους κανόνες ε, χρήσης ε, και την μελλοντική κείμενη νομοθεσία της Ένωσης, θα πρέπει να πηχούμε και την πραγματικότητα της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Δεύτερον, ε, οι Αρουμένοι ξέρουν πώς να προσαρμόζουν τα διάφορα συστήματα. Υπάρχουν και κατευθυντήρες γραμμές της ΙΑΤΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόζονται με συνέπεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ελπίζουμε να πιστούν όσοι δεν έχουν πιστεί ότι το 85-15 δεν αντιβαίνει στα συμφέροντά τους. Ε, κατά τη γνώμη μας ε, δεν συνεπάγεται αυτό αυξημένο λειτουργικό κόστος για τους αερομεταφορεί. Ε, και θα θέλαμε να επιληθείτε και εσείς του ζητήματος. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες άλλες παρατηρήσεις για τα νέα δίκτυα αερολιμένων. Νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί σύγχυση. Να κοιτάξουμε τις τροπολογίες αλλά υπό την προϋπόθεση επιτρέψτε μου να έχουμε ένα σύστημα για τα κράτη-μελή χειρισμού των δεδομένων, κυρίως για τις προθέσεις αεροπορικών δρομολογίων, για να έχουμε δυνατότητα συντονισμού, κυρίως σε περίπτωση κρίσης. Δηλαδή, ο συντονιστής του δικτύου, του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα παρέμβασης για τον προσδιορισμό των χρονοδιρίδων, ζητήματα ιδιοκτησίας κλπ μετά από όριμη σκέψη δεν ε, κρίνουμε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα χρήση. Έτσι ορίζεται στην πρότασή μα η χρονοθυρίδα. Για να ρυθμιστεί το ζήτημα, να πάει στιγμή, θα πρέπει ε, να ε, υπάγεται η χρήση στου κανόνε που εσεί θα έχετε θεσπίσει. Γιατί λύνεται και το δίλημα ποιο είναι ο ιδιοκτήτη σε σχέση τώρα με την εμπορία χρονοθυρίδων και τα ωφέλη, το κέρδος από αυτή την εμπορία. Ναι, είναι δελεαστική ιδέα, αλλά στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Τράν είχαμε προβλήματα ε, σε σχέση με την αποθάρρυνση ε, της εμπορίας στο δευτερογενή αγορά και άρα αποδυνάμωση αποτελεσματικότητας του νέου συστήματος. Ε, θα πρέπει να γίνεται η πληρωμή μέσω αεροπορικών τελών και όχι μέσω ενός μεσίτη χρονοθυρίδων. Για το τέλος κράτηση διαχείρισης όντως είναι ε, αποτελεσματικό εργαλείο προ ε, χρήση των αερολιμένων για να λυθούν σχετικά προβλήματα όπως το Düsseldorf που το έχουν δοκιμάσει πειραματικά και νομίζω ότι λειτουργήσε αισίω, διότι θεωρείται παράνομη η έξτρα χρέωση. Μπορούμε να ε, περιοριστούμε στην κλίμακα. Δεν χρειάζεται να ισχύει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω πρέπει να είναι ουδέτερη η νέα διάταξη ω προ το εισόδημα. Δηλαδή να μην κερδίζουν οι λεφτά από τους ε, αερομεταφορείς κατά αυτόν τον τρόπο οι αερολιμένες ε, γιατί δεν είναι περιορισμένη η ρευστότητα πλέον των αερομεταφορέων. Ζητώ συγγνώμη με ακρηγόρησε, αλλά ήθελα να σχολιάσω το θέμα των ε, χρονοθυρίδων και το 80-20 γιατί είναι ύψης τη σημασία. Ευχαριστούμε. Πριν ακούσουμε και πάλι τον κύριο Μπολντή να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει στους αερομεταφορείς μία επιστολή όπου αναφέρεται ε, αυτή η δυνατότητα 85-15 από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδέχεται να υπάρξουν αντίπεινα. Αντίπεινα λέει στην επιστολή. Μήπω ε, ξέρετε κάτι σχετικό πρωτού μπει στο συνολικό πακέτο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να, ε, τα, να παλέψω με του Αμερικανού, αλλά έχουμε 5-6 μάχε, προϊούσε μάχε. Α περιοριστούμε λίγο. Τι λέτε εσεί, κύριε Μπάλντεν. Ο αντιπρόεδρος Κάλλας πήρε ε, την επιστολή από την ε, ομόλογό του και φαντάζομαι ότι για αυτή την επιστολή μιλάτε από πλευρά τη αρχή ρύθμιση των ερωλημένων στη ΣΥΠΑ. Κοιτάξτε, ω απάντηση θα σα έλεγα ε, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, δεν Πρόκειται για ένα σύστημα εμπορίας όπως το ETS, δηλαδή αν ε, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να προσαρμόσουν τους κανόνες που προτείνει η ΆΤΑ, διότι εξάλλου οι Αμερικανοί δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες, ε, τους διεθνείς κανόνες. Ε, καλό θα ήταν με αυροφροσύνη να πούμε ότι με χαρά να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω, Πρόεδρε, ότι είναι ρεαλιστικό κακό αυτό το σενάριο ε, περί αντιπίνων. Ε, ευχαριστούμε, ο κύριος ε, Ούτζες. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο, γιατί κυρίως κατάλαβα και εκτίμησα την επικοδομητική και υπεύθυνη προσέγγιση που είχαν από πλευράς όλων των ομάδων και όλων των παρεμβενόντων ε, στην ε, σύνταξη της έκθεσης. Επίσης θα πρέπει να πω ότι εκτιμώ την ευελιξία που επιδεικνύει η Κομισιόν η οποία είναι ναι μεν σταθερή για ορισμένα, αλλά έχει αφήσει και κάποια ανοίγματα που πιστεύω θα πρέπει να τα δεχτούμε και να τα εκμεταλλευτούμε στη διατύπωση των συμβιβαστικών μας προτάσεων. Έτσι θα προχωρήσει καλά το θέμα μας. Δεν θέλω να σταθώ περισσότερο σε όλα αυτά, γιατί χρησιμοποίησα αρκετό χρόνο στην αρχή, όμως θα ήθελα να πω κάποια λόγια, κάποια πράγματα. Δεν ανέφερα, ας πούμε, το business aviation, γιατί είναι μια πτυχή που από τώρα, από, που εκφράζω την, το ανοιχτό μου πνεύμα, γιατί εξ αρχής πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα κομμάτια ε, ενέργειας κυκλοφορίας που είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε όντω να ολοκληρώσουμε το σύστημα των μεταφορών καθώς και το θέμα των ενσωματωμένων εισιτηρίων που, με το σύστημα το σιδηροδρομικό που βαίνει προς την οπτική που έχουμε συζητήσει άλλες φορές και όπου θεωρώ πως υπήρξε αρκετά γενική συμφωνία από πλευρά των διαφόρων συναδέλφων. Υπάρχουν τώρα κάποιες πτυχές που πρέπει να αποσαφηνίσουμε όπως το θέμα της συμβατότητας ανάμεσα στην επιλογή μας και την επιλογή των ε, εξωευρωπαϊκών αερολιμένων επί των οποίων θα εμβαθύνουμε σίγουρα πριν να φτάσουμε σε συμπέρασμα ώστε να μην μείνει ένα σύστημα ε, κουτσό και κλεισμένο στον εαυτό του, μέσα στο ευρωπαϊκό δηλαδή πλαίσιο μόνο, αλλά να μπορεί να και, συνδυαστεί και να ε, ε, συμφιλειωθεί με όλα τα συστήματα. Βέβαια, εμείς ως νομοθέτε θα πρέπει να αντιπροσωπεύσουμε με αξιοπρέπεια τα συμφέροντα για τα οποία αγωνιζόμαστε, που είναι κυρίως τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και τα συμφέροντα των θεσμών του οποίους εμείς εκπροσωπούμε. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά κήρυξη πολέμου, σημαίνει διαθεσιμότητα και διάλογο. Και σε αυτή τη γραμμή θέλω να διατηρήσω τη δράση μου και τη δράση από πλευράς των σκιωδών που μέχρι στιγμή συνεργάστηκαν καρποφόρα μαζί μου. Ευχαριστώ. Να θυμίσω στους ε, συναδελφούς πως η ψηφοφορία θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου. Θα περάσει κανονικά από την Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Με τα άλλα δύο κομμάτια αυτό που είναι γνωστό ως πακέτο των αεροδρομίων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ούτζες. Και έτσι ερχόμαστε στο τέλος της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών προγραμματισμένη για τις 5. Θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους πως η αυριανή συνεδρίαση γίνεται σε άλλη αίθουσα. Είναι στην αίθουσα Α3G3. Οπότε <clears throat> να πάρετε όλα σας τα χαρτιά μαζί. Και αύριο το πρωί θα τα πούμε στην Α3G3. Διακόπτουμε μέχρι τις 5 λοιπόν, όπου θα συναντηθούμε τους συντονιστές. Ευχαριστώ.